La Ξεκινάει η σύνοδος, συνεχίζεται η σύνοδος. Παρακαλώ καθίστε, έχουμε μια μεγάλη μέρα ψηφοφορίες και σήμερα θα προσπαθήσουμε να επιτελέσουμε το καθήκον μας όσο δυνατόν πιο ευχάριστα και γρήγορα. Να χαιρετήσω τον Μαρτίν Σουλτ, απερχόμενο πρόεδρο και να τον ευχαριστήσω για το έργο του σας εύχομαι, όπως έκανα και στη συνάντηση που είχαμε, ό,τι καλύτερο για την πολιτική σας διαδρομιά στη Γερμανία.